Okay, so now the com I think we have a quorum. Yes, we do. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Διαθέτουμε απαρτία. Ξεκινώ. Καλωσορίζοντάς σας στην συνάντηση της Επιτροπής Αναφορών. Να σας ξανακαλωσορίσω και στις Βρυξέλλες, όσοι φύγατε για τις διακοπές του Πάσχα. Ελπίζω να περάσετε καλά στις διακοπές σας δημιουργικά, να ξεκουραστήκατε, τουλάχιστον εγώ τα κατάφερα, έτσι ώστε να έχετε γυρίσει πίσω ανανεωμένοι και έτοιμοι να ασχίσετε τα καθήκοντά σα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ημερήσια μα διάταξη. Πρώτο, πρώτο θέμα, σημείο 2, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα απλώ να σα ενημερώσω ότι η ψηφοφορία για την έκθεση για τα παιδιά ε, θα γίνει στις 3 Μαΐου. Έχει αναβληθεί η κυρία Εύη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να λάβω τον λόγο για τόσο ακολούθησαν την τελική ψηφοφορία της ομάδας εργασίας που αφορά την καλομεταχείριση των ανηλίκων. Ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας θέλω να αναδείξω την προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας όλα όσα έγιναν επί πάνω από έναν χρόνο που κάτσαν οι εργασίες. Ήταν τα θέματα πολύ δύσκολα. Όλα τα θέματα που αφορούσαν την ζωή, τη μεταχείριση των ανηλίκων. Μια πολιτική ομάδα, η άλλη, κατέβασε 22 τροπολογίες που αφορούσαν την ακύρωση του τελικού εγγράφου. 22 παραγράφους. 12 από αυτές τις τροπολογίες απεσύρθησαν μόλις σήμερα και κατόπιν της ε, ψηφοφορίας που θα γίνει αύριο. Όλα αυτά, την παραμονή μα, την παραμονή της ψηφοφορίας. Πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, πρόκειται για κάποια απόφαση που θέλει να ακυρώσει όλο αυτό το έργο της ομάδας εργασίας. Αγνοεί όλες αυτές τις προσπάθειες η ομάδα των φιλελευθέρων. Όλα αυτά όσα κάναμε αυτή τη χρονιά. Ξέρω ότι όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να κατεβάσουν κάποια τροπολογία και την διατυπώνουν όπως νομίζουν ότι πρέπει. Αλλά νομίζω ότι είναι απογοητευτικό το ότι και η Πρόεδρος προσυπέγραψε αυτές τις τροπολογίες. Η Σεσίλια Βίξτρομ. Έτσι ακυρώνεται, έτσι απαξιώνεται το έργο της ε, ομάδας εργασίας μας. Το έργο των βουλευτών. Έτσι, μας αφαίρεται την νομιμοποίηση. Κάποιες τροπολογίες ως ε, προτάσεις εγκρίθηκαν και επιψηφίστηκαν και από την ίδια την άλλη. Και εγώ, όπου σαν πρόεδρος, πάντοτε λάμβανα υπόψη, ζήγιζα τις ευαισθησίες όλων των πολιτικών ομάδων. Πάντοτε ήμουν διαθέσιμη να αφουγκραστώ τις ανησυχίες τους. μέχρι την τελευταία συζήτηση που συζητήσαμε το σχέδιο εκειμένου και να σας πω δεν είχαμε ιδιαίτερε επικρίσεις από εσάς από την ομάδα ποτέ δεν ήρθατε στις εργασίες μας να παραστείτε να συμμετάσχετε Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προσβλητική αυτή η συμπεριφορά σας. Έτσι, αυτό το οποίο κάνετε αντιβαίνει και στο θεσμικό σας ρόλο. Και έτσι αμαυρώνεται και την εικόνα της Επιτροπής μας. Τώρα, εν κατακλείδη, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αντίθετα από άλλα έγγραφα εργασία των, ας πούμε, των επισκέψεων, των ε, αποστολών ε, των πραγμάτων, εμείς, σαν πάντα εργασία στο σώμα του κειμένου μας είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε τροπολογίες. Αυτό όμως συνήθως δεν συμβαίνει. Και εμείς το κάναμε αυτό γιατί προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε, να βρούμε σύγκληση απόψεων, να μπορέσουμε να συγκεράσουμε τη γνώμη της πλειοψηφία αν όχι την ομοφωνία. Εντάξει, αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει τελικώς. Επίσης, για τις ε, συστάσεις, τις προτάσεις. Έχουμε το πρώτο σχέδιο κειμένου το οποίο εγώ σας ε, παρουσίασα και προσπαθήσαμε επίσης να έχουμε και εδώ πολυφωνία, να συμμετάσχουν όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου και όλα αυτά, να τα φτιάξουν μια σύνθεση, έναν συμβασμό. Και η Άλντε για η κυρία Τούμ είπε όχι σε αυτή την προσέγγιση Οπότε, εγώ αυτό ως πρόεδρος επί πέντε μέρες σας να το δουλέψω, να κάνω τη σχετική πρόταση. Άλλωστε όλες οι ομάδες επί δύο εβδομάδες είχαν διάστημα και χρόνο να κατεβάσουν τις τροπολογίες τους. Εγώ δημοσία καταγγέλω αυτό το οποίο συνέβη. Αυτό θα πρέπει να λεφθεί υπόψη για το μέλλον, για να μην ξαναγίνει θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο μέλλον είναι αφόρητη μια τέτοια συμπεριφορά. Κυρίως από την πρόεδρο ο θεσμικός της ρόλος είναι να προσφέρει κάποιες εγγύησεις αξιοπρέπειας, αξιοπρέπειας διαφύλαξης της εικόνας της Επιτροπής των Αναφορών. Εγώ προσπάθησα να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο δημοκρατικά, με διαφάνεια, με πλουραλισμό, με ανοιχτό πνεύμα. Είμαι περήφανη για τον τρόπο που δουλέψαμε στην ομάδα εργασία και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετέσχουν. Είπαμε ότι αποσύρονται τι 12 τροπολογίε, αλλά θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει όσον αφορά το τελικό κείμενο τη ομάδα εργασία. Mrs. Tanoka. Thank you, Χαίρομαι που υποβάλλεται μια ε, λογική πρόταση για να λυθεί αυτή η πολύ περίεργη για εμένα κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω γιατί συμμετέχω στην Επιτροπή Αναφορών εδώ και πολλά χρόνια σε παλαιότερες διερευνητικές των πραγμάτων ε, αποστολές ε, είχαν υπάρξει κάποιες διαφωνίες αλλά πάντοτε το λύναμε τα προβλήματα και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί και αυτή τη φορά. Ε, οι τροπολογίες αρχικά του κ. Τρόβαλοφ και μετά η πρόταση που υπεκλήθη να αναβληθεί η ψηφοφορία Νομίζω ότι αν αναβληθεί η ψηφοφορία θα μας δοθεί η δυνατότητα να συναντηθούμε για να καταλάβουμε γιατί υπευλήθησαν αυτές οι 22 τροπολογίες. Οι περισσότερες τροπολογίες από αυτές ζητούν διαγραφή κειμένου και οποτεδήποτε προτινόταν ε, εναλλακτική διατύπωση, άλλο κείμενο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να πω ότι το νέο κείμενο ήταν καλύτερο. πολιτική μας ομάδα εκπροσωπήθηκε από την υποφαινόμενη σε αυτή την ομάδα εργασίας και οποτεδήποτε έλειπα ήταν παρουσία βοηθός μου δεν μπορώ να πω το ίδιο για την άλλη. Ε, Έλειπαν δηλαδή συχνά οι εκπρόσωποι της άλλη Και να βλέπω τώρα τροπολογία στις τελευταίες στιγμής ε, με εκπλήσει, με σοκάρει και ελπίζω όλα αυτά να οφείλονται σε μια παρεξήγηση εξαιτία τη έλλειψη χρόνου. Ίσως επειδή κάποιος δεν διάβασε προσεκτικά το κείμενο. Για να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτό που προτείνεται. Ξέρετε, μερικέ φορέ πολύ συχνά εμεί τα μέλη του Κοινοβουλίου βασιζόμαστε πολύ στου βοηθού μας και ίσως αυτό να μην είναι και τόσο καλή ιδέα πάντα. Ε, ε, η πρότασή μου είναι να αναβληθεί η ψηφοφορία, να γίνει μια ειλικρινή και πλήρη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Έχουμε μια παροιμία που λέει ότι τελικά το, ο σωστός λόγος, η λογική θα επικρατήσει. Σας ευχαριστώ. Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω την αναταραχή όταν το ζητούμενο είναι η καταθέση τροπολογιών Κάθε πολιτική ομάδα έχει το δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚ και του ΑΛΔΕ και η πρόεδρος μιας επιτροπής είναι επίσης ευρωβουλευτής που έχει το δικαίωμα να καταθέτει τροπολογίες οι οποίες ψηφίζονται. Είναι μια κανονική δημοκρατική διαδικασία. Αυτό ως προς το ένα. Ως προς το δύο το έχω απογραμμίσει δίπλο υπογραμμίσει, κάτι δεν λειτουργεί, μοιάζει να μην λειτουργεί. Επειδή αναβάλαμε την ψηφοφορία για την έκθεση, Και η συναδελφός είπε ότι θέλει να μιλήσουμε ειλικρινά. Εμείς στο ΕΛΚ το θέλουμε επίσης. Η συναδελφός Πιτέρα μας εκπροσώπησε στην ομάδα εργασίας και εκεί τη έλειπε αυτή η ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, επίση η ενασχόληση με τις προτάσεις των άλλων πολιτικών ομάδων. Και όταν η διάθεση συμβιβασμού δεν είναι ιδιαίτερη, τότε στο τέλος επέρχεται κατάρρευση. Εμείς ως πολιτική ομάδα δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, αλλά δεν προσπαθήσαμε ποτέ να το κρύψουμε. Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση αυτή, η οποία είναι μονόπλευρη η οποία χρήζει σίγουρα τροπολογιών και είμαι σίγουρος πως και άλλες πολιτικές ομάδες όπως η Άλντε έχουν καταθέσει τροπολογίες. Γι' αυτό και πρέπει να εκμεταλλευτούμε από την αναβολή της ψηφοφορίας για να βελτιώσουμε το κείμενο και αυτό είναι μια κανονική δημοκρατική διαδικασία και δεν υπάρχει κανένας άλλος στη λίστα μου επί του παρόντος. Συνάδελφοι, μια σημαντική αποσαφήνιση υπάρχει κάποια εκεί η κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Επίση και εγώ συμφωνώ με τους συνάδελφους ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση ειλικρινίας ε, και να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε. Ότι αυτές οι τροπολογίες ήρθαν πολύ πολύ τελευταία στιγμή, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, και την προέλευση των σκέψεων επίσης των τροπολογιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Ε, ε, στα πρότεινα να κάνουμε ένα προγραμματισμό από τώρα, σύντομο, πώς θα εξελιχθεί η πορεία της έκθεσης. Πότε θα γίνουν συζητήσεις, πότε θα ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες. Να μην τα αφήνουμε απλά έτσι το χρόνο και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. And that concludes... Σας ευχαριστούμε. Μπορούμε να πω ότι ολοκληρώσαμε το τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα σημεία της σημερινής της διάταξης, γιατί είναι παρόντες και ορισμένοι από τους προσφεύγοντες. Θα ήθελα, ήθελα να είμαι πλήρως ξεκάθαρη. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω δικαίωμα να εκφράζω τι πολιτικέ μου πεπιθήσει. Ωστόσο, ω πρόεδρο τη Επιτροπή έχω ιδιαίτερε ευθύνε, αρμοδιότητε. Αυτή τη στιγμή μια έκθεση, μια προφορική, ένα προφορικό ερώτημα έχει υποβληθεί θα, και θα την υποστηρίζω ε, μέχρι τελευταία ρανίδο, επειδή αυτό είναι ο ρόλο μου ω πρόεδρο τη Επιτροπή, ανεξαρτήτω εάν συμπίπτει με τι προσωπικέ μου πολιτικέ πεπιθήσει. Αυτό είναι ο ρόλος μου. Όμως αυτό ισχύει από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση της Επιτροπής. Μέχρι να φτάσουμε σε απόφαση της Επιτροπής έχω δικαίωμα να εκφράζω τις προσωπικές μου πεπιθήσει όπως οποιοδήποτε άλλο μέλος του Κοινοβουλίου. Αν ένα συνάδελφος μου ζητήσει να συνυπογράψω μια τροπολογία και συμφωνώ, το πράττω όπω οποιοδήποτε γιατί αν θεωρώ ότι συμπίπτει με την πολιτική μα γραμμή, τη γραμμή τη ομάδα μα, βεβαίω έχω το δικαίωμα να το πράξω. Τώρα, για ζητήματα παιδιών, ε, κράτηση παιδιών, ε, τα θέματα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ε, τα θεωρούν σημαντικά. Γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε και η ειδική ομάδα εργασία έτσι ώστε να γίνει μια συζήτηση περισσότερο σε βάθο μεταξύ των μελών. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε διάσταση απόψεων όσον αφορά την οργάνωση των εργασιών της ομάδας. Τη μεθοδολογία, τους, ο, τον που ε, καλέσαμε, ο οποίος δέχθηκε κριτική από μεμονωμένα μέλη και από ολοκλήρες πολιτικές ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κριτική εκφράστηκε με τρόπο ανοιχτό και ξεκάθαρο ε, προς όλους Μέρος αυτής της κριτικής είναι η υποβολή τροπολογιών προς το κείμενο της ε, ομάδας εργασίας. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό με αυτή τη διαδικασία, με αυτή τον τρόπο λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Γνωρίζω επίσης ότι η απόφαση για την αναβολή της συζήτησης ε, στην Επιτροπή του κειμένου ήταν ομόφωνη. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους κοιόδες εισηγητές να συναντηθούν άλλη μια φορά, προσπαθώντας να βρουν κάποιους συμβιβαστικές λύσεις για να καταλήξουν σε κείμενο το οποίο να καλύπτει τους πάντες. Ε, εγώ καλωσορίζω αυτή την απόφαση γιατί θεωρώ είναι προς το συμφέρον και το, το βέλτιστο συμφέρον της Επιτροπής. Ε, εγώ επίσης έχω ενημερωθεί ότι η σκιώδη τη έχει ζητήσει ε, συνάντηση των σκιωδών πριν από τι διακοπέ του Πάσχα και ότι ήταν διαθέσιμη να συναντηθεί και να, να, συναντηθεί και να συζητήσει με του συναδέλφου. Ελπίζω λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι να καταφέρετε να, να συναντηθείτε και να συζητήσετε έτσι ώστε η ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσει ομαλά. Δεν θα δώσω το λόγο πλέον για το θέμα αυτό σε κανέναν άλλον. Υπάρχουν άνθρωποι, ε, πολίτες που έχουν υποβάλει αναφορές και μας περιμένουν. Κυρία Εύη, δεν είναι δίκαιο αυτό κυρία Πρόεδρε. Αυτό που είπατε είναι απολύτως ε, λανθασμένο και απαράδεκτο. Είπατε ότι ασκήθηκε πολύ κριτική και ότι ασκήθηκε κριτική σε πολλούς από πολλά από τα πράγματα που έκανε η ομάδα εργασίας. Αυτό δεν ισχύει. Ένα μέλος μονάχα μίας πολιτικής ομάδας συστηματικά επέκρινε την, το έργο της ομάδας εργασίας. Ε, ζητώ συγγνώμη ε, το ΕΛΚ για πρώτη φορά δεν βρίσκεται με την πλειοψηφία. Μόνο αυτό συνέβη. Έχουμε δημοκρατία. Αυτό που συνέβη είναι ότι η πλειοψηφία της ομάδας εργασίας ελάμβανε τις αποφάσεις. Αυτό έγινε. Και, και μπορούν να με επιβεβαιώσουν όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας. Θα συμφωνήσουν νομίζω όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας ε, με ειλικρίνεια ότι έτσι έγιναν τα πράγματα αφού λέμε ότι μας ενδιαφέρει τόσο η ειλικρίνεια και το να μιλούμε ξεκάθαρα. Και ε, πρόεδρος, εντάξει, κάνατε τη διευκρίνηση, σας ζήτησε και κύριος... Όταν άρχισα να εργάζομαι στην ομάδα εργασίας αυτή, φυσικά και εκπροσωπούσα το ΕΛΚ αλλά αυτό ήταν δευτερεύον απέναντι στην ευζοία των παιδιών. Μιλήσαμε για μειοψηφίες, πλειοψηφίες. Το πρόβλημα όμως είναι πως το ΕΛΚ δεν επιζητεί να λύσει το πρόβλημα των παιδιών δεν είναι ένα δικαίωμα το οποίο υπερισχύει του άλλου. Δεν μιλούμε για μια πλειοψηφία ή μειοψηφία ψήφων. Το ζητούμενο είναι να επιτύχουμε με αποτελεσματικό τρόπο στόχους με την εργασία μας. Εμείς πιστεύουμε πως η έκθεση αυτή είναι μονόπλευρη. Όχι επειδή δεν συμπεριλήφθηκαν οι τροπολογίες μας, αλλά επειδή δεν λύνει το πρόβλημα που θέλαμε να λύσουμε εδώ. Είχαμε αμφιβολίες όσον αφορά τους ειδήμονες που συμμετείχαν στην εργασία. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό, αλλά θα, αλλά θα χρειαστεί να αναφέρω ξανά όλα τα επιχειρήματα. Έχω αμφιβολίες για την ποιότητα των πραγματονόμων αυτών. Ήταν πάντοτε συναισθηματικά φορτισμένοι από τις δικές τους εμπειρίες. Δεν ήταν πηγές αντικειμενικής ενημέρωσης και αντικειμενικές πηγές γνώσης. Το ζητούμενο ήταν η έκθεση αυτή να γίνει αντικειμενική. Θέλαμε κάτι αντικειμενικό, να επιτύχουμε ένα στόχο. Έτσι δεν είναι. Η κριτική αυτή την οποία που και που δέχθηκα εδώ, η κριτική αυτή δεν ήταν πολιτική, αλλά ρητορική. Εντάξει, συναδελφοί, ας προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Θα έχουμε μια ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, αυτό συμφωνήθηκε ήδη. Στοιχείο 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου έχουν διανεμηθεί, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούνται εγκεκριμένα. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση για τώρα και κάμια άλλη παρατήρηση στα διάφορα, οπότε περνούμε στην πρώτη σημερινή αναφορά, η οποία είναι η 1236 του 2015 του Μπρόνις Ροπέ, που φέρει 4.500 υπογραφές σχετικά με ανησυχίες με τον γαλακτοτομικό τομέα στη Λιθουανία. Ο αναφορέας δεν βρίσκεται εδώ. ο, αναφέρον, είχε ανακοινώσει πως θα βρισκόταν εδώ, αλλά καθώς δεν βρίσκεται εδώ, το λόγο έχει η εκπρόσωπος της Επιτρο... Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μισόν. Ελπίζω να είναι εδώ. Ναι, εδώ είμαι. Κύριε Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλους. Κύριε Μιζόν λέγομαι, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής ε, Πολιτικής στη Επιτροπή. Ο προσφεύγων στην αναφορά του αναφέρει ότι η τιμή του γάλακτος στη Λουθουανία είναι η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αποδίδει, εξηγεί αυτό με το ρωσικό εμπάργκο και ε, τις ε, επιδοτήσεις οι οποίες είναι μικρές κατά την άποψή του και εκφράζει τέσσερα αιτήματα. Να αυξηθεί η υποστήριξη προς τις χώρες εκείνες που έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο, ζητά να εγκριθεί νομοθεσία κατά των στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό, του του ανταγωνισμού μάλλον. Τρίτον, ζητάει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών. Και τέταρτον, ζητάει να υπάρξει ε, μια νέα, ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα γαλακτοκομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε προετοιμάσει μια γραπτή απάντηση, ε, την οποία σα υποβάλαμε το προηγούμενο καλοκαίρι και στην οποία ε, Αναγνωρίζουμε ότι η Λιθουανία έχει πληγεί ιδιαίτερα από το ρωσικό εμπάργκο και αναφέρουμε ότι το γεγονό αυτό έχει ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κατέρτισε τα διάφορα ε, μέτρα στήριξης των παραγωγών από το 2014. Υπήρξαν στοχευμένα μέτρη, μέτρα υπέρ των γαλακτοπαραγωγών στα βαλτικά κράτη, ανάμεσά τους και η Λουθανία, ε, μετά και υπέρ των παραγωγών στην Φινλανδία, δηλαδή τα τρία βαλτικά κράτη και η Φινλανδία ήταν αυτές που ε, κυρίως επλήγησαν. Μετά το 2015 και μετά το 2016 ε, συμπεριλάβαμε, μάλλον υιοθετήσαμε και άλλα μέτρα στήριξης, επιπλέον χρήματα, τα οποία όμως αφορούσαν και τα 28 κράτη-μέλη. Ωστόσο, όταν έγιναν οι υπολογισμοί για να προσδιοριστούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε χώρα, ε, λάβαμε υπόψη το ρωσικό εμπάργκο και το γεγονό ότι έχει ιδιαίτερα πλήξει τη Λιθουανία και αυτό οδήγησε στο, τα, τα χρήματα που ήταν διαθέσιμα για τη Λιθουανία να είναι αυξημένα. Επομένω, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αυτά τα μέτρα και τα έλαβε πρόσφατα. Ε, χρήσιμο θα ήταν επίση να υπενθυμίσει κανείς ότι οι άμεσε ενισχύσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ΚΑΠ και υπάρχουν και άλλες πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και γενικότερα για τη γεωργία αλλά και πιο συγκεκριμένα για τον ε, τομέα των ε, γαλακτοκομικών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μαριά. Πρόεδρε, εγώ θα πάρω αφορμή από αυτή την αναφορά, διότι το ζήτημα των επιπτώσεων του ρωσικού εμπάργου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και φυσικά αναφέρθηκε ότι υπήρξαν συγκεκριμένες χώρες οι οποίες επλήγησαν. Να επιστημάνω ότι από τα μέτρα για το ρωσικό εμπάργο έχει πληγεί και η ελληνική αγροτική οικονομία και η κτηνοτροφία. Και αυτά που δόθηκαν ουσιαστικά ως αποζημιώσεις είναι ψίχουλα. Ε, είχα κάνει μια ερώτηση έγκαιρα όταν ε, ε, επευλήθησαν το, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τα αντίμετρα από την πλευρά της Ρωσίας μαζί με συναδέλφους από την Ιταλία για το τι θα υπάρξει ως αποζημίωση για τους Έλληνες αγρότες, τους Ιταλούς αγρότες και φυσικά τους κτηνοτρόφους. Νομίζω ότι μετά από πολλές συζητήσεις τα μέτρα τα οποία υπάρχουν και για τους κτηνοτρόφους δεν είναι αρκετά και φυσικά θεωρώ ότι η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια σε ένα πολιτικό ζήτημα η απόφαση τι θα γίνει με, το, τα μέτρα κατά της Ρωσίας. Εγώ επιμένω ότι πρέπει αυτά να αρθούν διότι δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την αγροτική οικονομία στην Ελλάδα και άλλες χώρες. Αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο θα αποφασιστεί σε άλλο επίπεδο. Το θέμα είναι να υπάρξει μια δίκαιη αποζημίωση όσων πλήττονται. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει ειδικότερα και με τις πολιτικές για το γάλα. Ε, πολιτικές στις οποίες θα αναφερθώ αργότερα γιατί υπάρχει επόμενη ε, αναφορά η οποία νομίζω επίσης έχει άμεση σχέση με τις τιμές του γάλακτος και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Ευχαριστώ. συμφωνούμε πως το ρωσικό εμπάργο έχει επιπτώσεις στη γεωργία και η χώρα μας πλήττεται στην Ευρώπη. Έχουμε και την κρίση του γάλακτος, η οποία δεν οφείλεται μόνο στο ρωσικό εμπάργο. Φυσικά και πρέπει να είμαστε δίκαιοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία γνωρίζει το πρόβλημα. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα και έκανε ό,τι μπορούσε. Δύο παραδείγματα μόνο γι' αυτό. Είχαμε τη δέσμη μέτρων, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε πως αν τα κράτη-μέλη δεν διατίθενται να καταβάλουν περισσότερα χρήματα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει τις δυνατότητές της να εξαντλούνται σε κάποια στιγμή. Και φυσικά όταν ένας τομέας παίρνει περισσότερα χρήματα, τα χρήματα αυτά αφαιρούνται από κάποιον άλλο τομέα. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που χρηματοδοτήθηκε εκτός προϋπολογισμού το ζήτημα του γάλακτος. Αλλά πρέπει να πούμε πως δεν έχουμε και πολλά περισσότερα χρήματα. Και θα χαιρόμουν πολύ εάν δεσμεύονταν και τα κράτη-μέλη, τα οποία με την καρδιά τους είναι από την πλευρά μας. Αλλά όταν το ζητούμενο είναι να πληρώσουν χρήματα, τότε συνήθως δεν είναι πια στο πλάι μας. Γι' αυτό και πιστεύω πως η αναφορά πρέπει να κλείσει. Οι δέσμες μέτρων είχαν λίγη ωφέλεια. Το ρωσικό εμπάργο, ναι γι' αυτό μπορούμε φυσικά να κάνουμε ένα πολιτικό ψήφισμα, είναι καθήκον όλων μας. Ισχύει και για τις δύο πλευρές να έχουμε ορθές σχέσεις με τη Ρωσία. Αν αυτές βασίζονται, βρίσκονται σε εταιρικό επίπεδο, τότε θα αποφεληθούν και οι δύο. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε αρνητικέ οικονομικές επιπτώσεις και από τις δύο πλευρές. Θα ήθελα όμως να καταγραφεί στα πρακτικά πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα άμεσες ενισχύσεις, παρεμβάσεις κτλ. Αυτό ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά. Δηλαδή συνοπτικά η αναφορά θα μπορούσε να κλείσει σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος στη λίστα ομιλητών. Οπότε πιστεύω πως μπορώ να προκαταλάβω τι, τι θα πει η Επιτροπή. Ακριβώς αυτό που είπε ο Πέτερ Γιάρ. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάρτησε οτιδήποτε δυνατόν. Και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε την αναφορά και να τη στείλουμε στις λιθωνικές αρχές για την ενημέρωσή τους, για να μάθουν πως υπήρξε μία αναφορά με πολλά την οποία αναφορά υποστήριζαν πολλοί πολίτες και για να επιστήσουμε την προσοχή των λιθωνικών αρχών στην αναφορά αυτή. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι υπέροχα. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η αναφορά 0967 του 2016 από τον Detlef Velbrock εκ μέρους της τοπικής αρχής του Λόκστετ σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των χαμηλών τιμών του γάλακτος στις γραφτοκομικές επιχειρήσεις της περιοχής. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ, οπότε πάλι δίνει το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, την κυρία Μισόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αναφορά αυτή, ο κύριος Φέλπροκ τονίζει το γεγονό ότι οι χαμηλές τιμές του γάλακτος δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτό οδηγεί σε αλλαγή στο, στη δομή της αγροτικής, ε, των αγροτικών περιφερειών ε, στα χωριά και ζητά αυτό να αντιμετωπιστεί σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση ζητά, αν ε, μάλλον αναφέρει, ότι αυτή η μείωση των τιμών στην πραγματικότητα δεν περνάει στον τελικό καταναλωτή. Οι καταναλωτέ πληρώνουν πιο ακριβά το γάλα του, ενώ οι μεγάλε επιχειρήσει διανομή είναι αυτέ που αυξάνουν τα κέρδη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι στον τομέα τη ρύθμιση των γαλακτοκομικών υπάρχουν και ευκαιρίε, υπάρχουν και προβλήματα. όπω γνωρίζετε, 29 δισεκατομμύρια ε, ευρώ είναι το ύψος της ε, ΚΑΠ, όχι μόνο άμεση ενισχύσει, αλλά εδώ συμπεριλαμβάνω και άλλα προγράμματα, όπω προγράμματα αγροτική ανάπτυξη και επίση ε, προγράμματα κοινή οργάνωση αγορά. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους βασικούς πυλώνες έχουμε και την πολιτική για την ποιότητα με την οποία προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την τοπική παραγωγή Υπάρχει επίσης και το λεγόμενο δίχτυ ασφαλείας, το οποίο συμπεριλαμβάνει μέτρα ε, ενίσχυσης κρατικής ε, ή αποθήκευσης προϊόντων. Ε, υπάρχουν και άλλα μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για να αντιμετωπίσουν προβλήματα ε, ταμιακής ρευστότητας, στοχευμένη βοήθεια σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να ε, βελτιωθεί, να, σταθεροποιηθεί η αγορά. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν, διάφορες, έχουν εκτός των άλλων ε, δυνατότητες ε, να αξιοποιήσουν τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτών επίσης. Υπάρχει επίσης και η πολιτική προώθηση των προϊόντων για να προωθούνται τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά σε τρίτες χώρες και υπάρχει και μια ομάδα εργασία για τις, την αγροτική παραγωγή, ε, η οποία συνεδρίασε καθ' όλη τη διάρκεια του 2016 με στόχο να δει πιο μακροπρόθεσμα τι πρέπει να γίνει και η οποία κατέληξε σε μια σειρά ε, συστάσεων, τις οποίες εξετάζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έγινε παράλληλα με το πρόγραμμα που είχε ήδη ξεκινήσει για, την προ... μια πρόταση εξυγχρονισμού της ΚΑΠ. Της... Με... Ορίζονται την επόμενη ΚΑΠ. Είναι μια διαβούλευση η οποία είναι ανοιχτή σε όλους ε, και στην οποία ζητούμε από όλους τους πολίτες να συνεισφέρουν. Ε, με προτάσεις έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί τη νέα ΚΑΠ. Ένα από τα ερωτήματα που έχει τεθεί σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, θα σας αναφέρω μάλλον μερικά, ζητούμε από τους πολίτες να μας πούν εάν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν κάπως περισσότερο για τα αγροτικά προϊόντα Πέρα από αυτά υπάρχει και το πακέτο γάλα, το για το γάλα, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους παραγωγούς να βελτιώσουν την διαπραγματευτική τους θέση στην ε, αλυσίδα την εμπορική. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια, υπάρχουν πολλά και διάφορα εργαλεία τα οποία δίνουμε στους παραγωγούς για να βελτιώσουν τη θέση τους και να εξασφαλίσουμε το μέλλον τους. Σα ευχαριστώ. Η πρόεδρος, εμεί σα ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει... Όχι, ο κύριο Μαριά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά αυτή η αναφορά θέτει πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και είναι ευκαιρία να τα θέσουμε εδώ. Βέβαια δεν έχουμε πάρα πολλού συναδέλφου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το ζήτημα της, πολιτικής, ε, της κοινής αγροτικής πολιτικής, διότι αυτό που εγώ τουλάχιστον θεωρούσα σημαντικό είναι ότι η βασική αρχή είναι η αρχή της κοινοτικής προτίμησης. Μόνο στη βάση αυτή μπορεί κανείς να δει μια σοβαρή ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι μια απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, μια συνεχή εισαγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να ε, υποβαθμίζεται το γεωργικό εισόδημα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα διαφοράς ως προς τα εργαλεία και την αρχή με την οποία ενεργούμε. Διαφωνώ με την πολιτική που έχει η Κομισιόν, το έχω πει αρκετές φορές και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το ξαναδούμε. Δεύτερο, σε σχέση με τα, ε, την ποιότητα, που είπαμε ότι η ποιότητα βασικά έχει σχέση με τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Βλέπουμε ότι αυτά πλήττονται και έχουν ε, πληγεί και από την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μεσημβρινής Αφρικής σε σχέση με την ΦΕΤΑ αλλά και με την ΣΕΤΑ διότι η ΣΕΤΑ πραγματικά έχει διαλύσει όλη, θα διαλύσει μάλλον την προστασία της ΦΕΤΑ ως προϊόν ονομασίας προέλευσης. Σας λέω ότι ήταν σοβαρό θέμα. Ήδη έχουν γίνει πολλές μεγάλες συγκεντρώσεις κτηνοτρόφων στην Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στον Τύρναβο και στον Αλμυρό αγροτικές κτηνοτροφικές περιοχές σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Η τιμή του γάλακτος, ιδίως του πρόβιου και του κατσικίσου, έχει πέσει πλέον, διότι δεν θα υπάρχει αυτή η προστασία στο προϊόν ονομασίας προέλευσης. Επισημαίνουμε ότι εγώ τουλάχιστον καταψήφισα τη ΣΕΤΑ και ένας από τους λόγους ήταν το ότι δεν προστατεύεται πλέον η ΦΕΤΑ ως προστασία ονομασίας προέλευσης για τον απλό λόγο ότι επιτρέπεται η παραγωγή φέτας μαϊμού, δηλαδή φέτας από αγελαδινό γάλα στον Καναδά και αυτό θα ανοίξει το δρόμο στην πορεία και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάψει αυτή η προστασία. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική στο θέμα αυτό η Κομισιόν, πρέπει να δει σοβαρά τα αιτήματα των Ελλήνων κτηνοτρόφων και μεταφέρω την αγωνία των Ελλήνων κτηνοτρόφων στο ζήτημα αυτό. Τρίτο θέμα, επειδή είναι εδώ η Κομισιόν για να τα ακούσει, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις κατασχέσεις που γίνεται στο εισόδημα των αγροτών. Δηλαδή οι αγροτικές επιδοτήσεις, οι επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων κατάσχονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ε, υπάρχει μια νομοθεσία που πέρασε από την Τρόικα και ως εκ τούτου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βλέπουν να έρχονται οι εισοδηματικές ενισχύσεις στο λογαριασμό τους αλλά μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται το κατάσχει το κράτο, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζε, οι ιδιώτε κλπ. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Τέταρτο ζήτημα είναι ότι πράγματι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική προστασία και για τον αγροτικό τομέα και ιδίω για του κτηνοτρόφου. Να σα πω λοιπόν, και το λέω στην Κομισιόν για να τα ακούσει, γιατί είναι εδώ, ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με του βοσκοτόπου. Διότι όταν μειώνονται οι εκτάσει των βοσκοτόπων, είναι προφανέ ότι και οι επιδοτήσει μειώνονται. Και σήμερα στην Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό, να σα ενημερώσω ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με του δασικού χάρτε. Χτε ήμουν δασικού χάρτε, δηλαδή τι είναι δάσο και τι δεν είναι δάσο. Ήμουν χτε ε, στην Καριστία, νότιο Καριστία, δηλαδή στην περιοχή τη Εύβοια, όπου το κράτος, το ελληνικό, με τις αποφάσεις που έχει πάρει, θεωρεί πολλές ιδιωτικέ εκτάσει, πολύ μεγάλε, και εκτάσει που ήταν βοσκότοποι, ως κρατικές εκτάσεις, ότι δήθεν ήταν παλιά δάσος και επομένως το κράτος θα πάρει πλέον αυτές τις ιδιοκτησίες και δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε οι κτηνοτρόφοι να ε, βόσκουν εκεί τα δικά τους ε, ζώα, κυρίως πρόβατα και κατσίκια. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα το φέρω με ερώτηση στην Κομισιόν. Θα ήθελα να το ακούσουν από πλευρά Κομισιόν γιατί είναι σοβαρό ζήτημα. Είναι μια εφαρπαγή της ιδιοκτησίας στην ουσία των Ελλήνων πολιτών προκειμένου να μετατραπούν σε δίθεν κρατικές γεές και εν συνεχεία να μπουν αυτά, αυτές οι μεγάλες εκτάσεις να περάσουν στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή στο ταμείο το οποίο προωθεί, προωθούν οι δανειστές για εκποίηση της δημόσιας περιουσίας ή να μπουν ως υποθήκη. Αυτά λοιπόν είναι σοβαρά θέματα. Είναι ευκαιρία το ότι τίθενται εδώ με αναφορές από άλλα κράτη, αλλά το θέμα της προστασίας των ε, ε, εκτινοτρόφων συνολικά και των Ελλήνων εκτινοτρόφων και αγροτών ειδικότερα, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να εκθέσω τα θέματα αυτά, να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι, να τα ακούσει και η Κομισιόν, διότι χθε πήρα μια δέσμευση μιλώντα στην Κάριστο απέναντι στου κτηνοτρόφου ότι αυτά τα θέματα θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει ενημέρωση και να υπάρξει και απάντηση από πλευρά Κομισιόν. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Αλλά υπάρχει όχι μόνο φέτα, υπάρχει και σαγκανάκι και, και χαλούμι και τα λοιπά. Η φέτα είναι η ναυαρχίδα <laughs> της ε, ελληνικής κτηνοτροφίας και θα πρέπει να προστατευτεί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, το ξέρω. Λοιπόν, να προχωρούμε. Πέτερ the floor is to you. Äh, Μην με παρανοήσετε, αλλά οι τιμές γάλακτος που καταβάλλονταν το 2016 δεν ήταν μόνο επικίνδυνα χαμηλές, αλλά ήταν μια ανέδεια ως προς, όσον αφορά την εργασία των γεωργών. Είναι γεγονός αυτό η Κομισιόν προσπάθησε να αντιδράσει και έχουμε συνείδηση του ότι ο γαλακτοκομικός τομέας ασκεί μεγάλη επιρροή στον γεωργικό τομέα γενικότερα και στη λειτουργία της υπαίθρου στο σύνολό της. Αλλά δεν πρέπει να υπερκαταπονήσουμε την Επιτροπή Αναφορών. Επί του, παρόντος έχουμε τη λεγόμενη διαδικασία Omnibus στο πλαίσιο της οποίας μπορούμε να επιτύχουμε μικρές τροποποιήσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα το ανέφερα αυτό στους αναφέροντες για το πώς θα συνεχιστεί μετά το 2020 η κοινή γεωργική πολιτική. Και στον γαλακτοκομικό τομέα πρέπει να διαπιστώσουμε πως απομένουν πολλά που πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε ισότιμους όρους, ισότιμα όπλα θα έλεγα, μεταξύ των αλυσίδων της αγοράς και των γεωργών αλλά πρέπει να αλλάξουμε μερικά όσον αφορά τις συμβατικές, τους συμβατικούς όρους επειδή εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγουμε περισσότερα γαλακτοκομικά από αυτά που εισάγουμε. Αυτό σημαίνει πως δρούμε σε μια παγκόσμια αγορά και πρέπει να φέρουμε σε μια ισορροπία την προσφορά και τη ζήτηση, ακόμη και αν η ζήτηση κυμαίνεται. Όλα αυτά τα συζητούμε. Θα έλεγα πως η Επιτροπή Αναφορών ως τέτοια μπορεί να κλείσει την αναφορά υποδεικνύοντας τις δραστηριότητες του και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της κοινή αγρογεωργικής περιοχής, πολιτικής συγγνώμη. Αλλά αυτό που απογοητεύει ως ειδικευμένος πολιτικός είναι οι τιμές αυτές οι οποίες ήταν γελίες για τον τομέα αυτό και ήταν η κήρυξη πολέμου ενάντια σε ένα ολόκληρο τομέα. Από τα χρήματα αυτά δεν μπορεί να ζήσει κανείς γεωργός. Ούτε μπορεί να επιβιώσει η ύπεθρος. Γι' αυτό και ήταν απειλητική η εξέλιξη αυτή, γι' αυτό και η Επιτροπή Αναφορών και η Κομισιόν ασχολήθηκαν τόσο εντατικά με το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Δεν έχω κάποιον άλλο στον κατάλογο ομιλητών. Οπότε πιστεύω πως μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Η πρότασή μου είναι να κλείσουμε την αναφορά σύμφωνα με αυτά που μάθαμε από την Κομισιόν καθώς ο αναφορέας προσκλήθηκε να σχολιάσει, να υποβάλει σχόλια στην διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης και αρνήθηκε ή μάλλον αμέλησε να το κάνει, γι' αυτό πιστεύω πως μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά αυτή και ρωτώ τους συναδέλφους μπορούμε. Το παίρνω ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ας πέρασουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το οποίο σχετίζεται με το ίδιο θέμα. Αναφορά 1199 του 2016 του Γερκ Πράλ σχετικά με την απόρριψη αίτησης ενίσχυσης για τη μείωση παραγωγής γάλακτος. Δεν βρίσκεται εδώ. Αλλά η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ και έτοιμη να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ε, κύριος Πράλ είναι αγρότης. Έχει περίπου 30 γαλακτοφόρες αγελάδες. Ήθελε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της μείωσης της παραγωγής. Αυτό το οποίο απεφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των μέτρων του Ιουλίου του 2016. Και η αίτησή του απερίφθη. Διότι ο κύριος Πράλ δεν ε, παραδίδει γάλα τον ε, Ιούλιο. Οργανώνει έτσι τη δουλειά του που σταματά την άνοιξη να παραδίδει το γάλα. Γεννούν οι αγελάδες το καλοκαίρι οπότε και τότε το σύνολο του γάλακτος το δίνει στα μοσχαράκια οπότε δεν έχει αποδείξει ότι παρέδωσε τον Ιούλιο του 16 γάλα. Οπότε θεωρεί ότι αυτό είναι δυσμενή διάκριση ει βάρο του, ότι είναι ζημία ει βάρο του, γιατί δεν μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή απήντησε εγγραφο ε, στην αίτησή του και για να καταλάβετε καλύτερα θα πρέπει να ξαναδούμε το γιατί ε, θεσπίσουμε αυτό το πρόγραμμα μείωση της παραγωγής. Το καλοκαίρι του 2016 ο κύριος ε, Γιάρτο ετώνησε πριν σωστά ότι υπήρξε κάποιο είδου ε, μείωση των τιμών στο γάλα. Οπότε με το που πήγαν τόσο χαμηλά οι τιμές, ε, ήταν, ε, ο λόγος που έγινε αυτό ήταν γιατί υπήρχε ανισορροπία ζήτηση και προσφορά. Οπότε είπαμε εμεί η ισορροπία θα επανέλθει εάν κάνουμε κάτι για την προσφορά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάσισε για αυτό το πρόγραμμα το οποίο πρόσφερε κάποια ευρώ για 100 ε, κιλά που δεν θα παρήγονται, για κάθε 100 κιλά που θα παρήγονται, σε όλου του παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το θέλανε. Οπότε ήταν ε, κούσια η συμμετοχή. Αλλά ε, η προπόθεση ήταν ότι θα έπρεπε να είναι ενεργή αυτή η παραγωγή για να είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα στην αγορά. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο υπήρξε μείωση στην παραγωγή. Να ξαναφέρουμε επομένω τις τιμές προς τα πάνω και τα πιο πρόσφατα δεδομένα ε, υπάρχουν για να δούμε κατά πόσον αν κάποιος δηλαδή παραγωγός είναι ενεργός και είπαμε ότι αυτό το, το κριτήριο θα ήταν εάν έχει δώσει ε, γάλα τον Ιούλιο. Και υπάρχει μια ρήτρα που λέει ότι αν κάνει επιλέξιμο στα πλαίσια του κοινωνικού κανονισμού, ο παραγωγό θα πρέπει να αποδείξει ότι παρέδωσε γάλα ε, τον Ιούλιο του 2016. Ο κύριος Πραλ δεν ε, πληρούσε τα κριτήρια της επιλεξιμότητας, οπότε δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Επομένως δεν είναι πρόκειτο για κάποιο είδου ε, ζημία που του επιφέραμε. Τώρα υπήρχαν και άλλα μέτρα τα οποία προεβλέπονται σε αυτό το πακέτο του Ιουλίου του 2016. Υπήρξε ένα μέτρο που νόμιτρο διανομής 50 ε, εκατομμυρίων ευρώ σε όλα τα κράτη-μέλη που δεν ε, συνεδέονται με κάποιο είδου ε, κριτήρια επιλεξιμότητας. Οπότε, για την ενημέρωσή σας, σας λέω ότι τώρα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Τώρα, επομένως, ε, βλέπουμε ότι η πρώτη χρήση του προγράμματος είναι η Γερμανία. Από πλώστορα της ε, υλοποίησης εφαρμογής όσον αφορά τη μείωση της παραγωγής, περισσότερο ωφελήθηκε από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα η Γερμανία. Και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ναι, εμείς ευχαριστούμε. Ποιος ο θέλει το λόγο. Γεια. Οι όροι είναι αυτοί που είναι και η κομισιόν. Πού θα το πω διαμόρφωσε το πρόγραμμα παραγωγή γάλακτο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τον Ιούλιο του 2016 έπρεπε να παραδώσει κανεί γάλα σε γαλακτοκομικέ μονάδε. Το γάλα δεν παραδίδονταν εκεί στι μονάδε αυτέ, Οπότε ο αναφέρον δεν δικαιούται ενίσχυση, Οπότε μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά και να το αποδείξουμε τα εθνικά προγράμματα στήριξης Λυπούμε γι' αυτό, αλλά είναι μονοσήμαντες οι προϋποθέσεις που καθόρισε η Κομισιόν. Τον Ιούνιο του 2016 έπρεπε να είναι κανείς παρα... γαλακτοπαραγωγός κάποιος για να λάβει την ενίσχυση αυτή και όχι άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το γάλα για τους μόσχους. Λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά κανόνε του παιχνιδιού πρέπει να καθοριστούν και υπάρχουν πάντα αυτοί που μπαίνουν έξω από τους κανόνες. Λυπούμε γι' αυτό, αλλά τότε ο αναφέρον πρέπει να αποταθεί στις, στα εθνικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Θα το κάνουμε ως εξής. Θα ακολουθήσουμε την πολύ σοφή συμβουλή του Πέτερ θα γράψουμε μία επιστολή στον αναφέροντα προτρέποντας τον να απευθυνθεί στις εθνικές αρχές για να αποφεληθεί από τα εθνικά προγράμματα στήριξης που διατίθενται. Και θα το κάνουμε με έναν πολύ συμπαθητικό τρόπο. Θα του στείλουμε μία επιστολή και θα του εκφράσουμε τη συμπάθειά μας για τη θέση του και θα του πούμε να έχει κατά νου πως υπάρχει μία εκκρεμούσα περίπτωση στο δικαστήριο αλλά πως αυτό δεν σχετίζεται με εμάς, με το πώς μεταχειριζόμαστε την αναφορά. Είναι μια εθνική δικαστική υπόθεση. Οπότε του στέλνουμε την επιστολή αυτή και μετά κλείνουμε την αναφορά, εντάξει. Η επόμενη, η 392 του 2015 του ή ΠΙΕΣ, εκ της Βρετανικής εκ μέρους της οργάνωσης Compassion in World Farming με υπογραφές από από που προωθούν την ορθή μεταχείριση των ζώων σχετικά με την ορθή μεταχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Ο κύριος Στίβενσον είναι εδώ και τον καλωσορίζω. Χαιρόμαστε πολύ για την εισήγησή σας. Σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε ελεγχούς για την ορθή μεταχείριση των αγελάδων σε πέντε κράτη-μέλη. Τα αποτελέσματα είναι ανα, αναμεικτά. Υπάρχουν θετικά ευρήματα αλλά και κάποιες ανησυχητικές πτυχές. Παραδείγματο χάρη στην Πολωνία η έκθεση δείχνει πως κάποιες αγελάδες εξωθούνται σε τόσο υψηλές αποδόσεις σε γάλα που το 1 τρίτο τους πρέπει να σφαγεί πρόωρα κάθε χρόνο. Στην η Ιρλανδία το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κοπή της ουράς των αγελάδων. Στην Αυστρία το 45-50% των αγελάδων είναι δεμένες σε κλειστούς χώρους για το περισσότερο του έτους. Στην, Εσθανο, στην Εσθονία η αναφορά αποκαλύπτει ειδήματα, κοψίματα, τραυματισμούς, μαστίτιδα και χολότητα. Η έκθεση σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων καταρτίστηκε από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών. Σύμφωνα με αυτήν, η ορθή μεταχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής είναι ίσως το, το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα μεταχείρισης των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης αναφέρει πως οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής που παράγουν μεγάλες ποσότητες γάλακτος έχουν υψηλά επίπεδα διαταραχών των άκρων, μαστίτιδας και αναπαραγωγικών διαταραχών. Η έκθεση της Επιτροπής τόνισε πως η αναλογία των αγελάδων που πλήττονται από μία ή περισσότερες από τις διαταραχές αυτές είναι υψηλή και πως τα ζώα ζουν σε κακές συνθήκες για ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους. Εμείς επισκεφτήκαμε 52 εκμεταλλεύσεις αγελάδων στη Γερμανία, τη Δανία και την Ισπανία το 2012. Βρήκαμε πως σε πάνω από 50% των εκμεταλλεύσεων που επισκεφτήκαμε, οι αγελάδες ήταν κλεισμένες σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο, όχι μόνο το χειμώνα, αλλά επίσης κατά την αυξητική περίοδο του χώρου του. Σε κάποια κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας, πολλές αγελάδες είναι δεμένες σε εσωτερικούς χώρους για σχεδόν όλο το χρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα 24 ώρες την ημέρα, όλο το έτος. Τα ζώα αυτά ούτε που μπορούν να κινούνται. Μπορούν να πάνε να ξαπλώσουν, να σηκωθούν και να κάνουν μερικά βήματα προς τα πίσω, προς τα μπροστά ή και πλάγια. Οι σημερινές αγελάδες εκτρέφονται για πολύ υψηλές αποδόσεις σε γάλα. Αλλά η μακροχρόνια γενετική επιλογή είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που προκαλεί κακές συνθήκες διαβίωσης και ιδίω προβλήματα υγείας σε αγελάδε γαλακτοπαραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, αναφέρει πως έχουμε 20 έως 25% χολότητα, το οποίο σημαίνει ότι 20 έως 25% των ζώων είναι χολά η ΕΦΣΑ αναφέρει πως δεν έχει επιτευχθεί κάποια μίεση στον επιπολασμό της χολότητα τα τελευταία 20 χρόνια και πω οι περισσότερες χολέ αγελάδε πονούν. Οι συνθήκε. Διαβίωση είναι συχνά κακέ. Οι αγελάδες βρίσκονται συχνά υπό συνθήκε συνοστισμού και έλλειψη καθαριότητα σε διαμερίσματα εκλοβού. Τα πατώματα είναι συχνά σκληρά και άβολα και οι κλοβοί, τα διαμερίσματα συχνά δεν έχουν σανό, άμμο ή κάποια άλλη στρώμη, το οποίο προκαλεί πληγές και βλάβες στα ζώα. Όσον αφορά την νομική κατάσταση, δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία ειδική για τις αγελάδες, οπότε πρέπει να βασιστούμε στην γενική οδηγία περί εκτρεφόμενων ζώων που ισχύει για όλα τα ζώα. Σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν πως οι εκτροφείς πρέπει να πάρουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν την ορθή μεταχείριση των ζώων και πως αυτά δεν εκτίθενται σε πόνο, δεν υποφέρουν ή δεν τραυματίζονται. Προτρέπουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσει την αναφορά ανοιχτή και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή καθοδήγηση στα κράτη-μέλη για τον τομέα των γαλακτοκομικών τους, καθορίζοντας τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες για να συμμορφωθούν με την γενική οδηγία και ιδίως με το άρθρο 3 αναφερόμενοι συγκεκριμένα στην αλαχιστοποίηση της χολότητας και της μαστίτιδας, στην αλαχιστοποίηση των τραυματισμών των, και των ειδημάτων και των βλαβών, πώς μπορεί να επιτευχθεί μια καλή σωματική κατάσταση. Ε, είδατε στις φωτογραφίες κάποιες πολύ λεπτές αγελάδες. Πώς μπορεί να, διασφαλιστεί, να διασφαλιστούν οι καθαρές συνθήκες εκτροφής για να μην πάθουν οι αγελάδες μαστίτιδα πώς μπορούν να διασφαλιστούν οι σωστές διαστάσεις των κλοβών, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η πρόσβαση των αγελάδων σε βοσκότοπους κατά την αυξητική περίοδο του χόρτου και πώς μπορεί να τερματιστεί αυτή η απέσια συνήθεια της πρόσδεσης των αγελάδων. Επίσης, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που απορρέουν από την εκτροφή για υψηλές αποδόσεις γάλα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ξεκάθαρη καθοδήγηση. Τι χρειά... Δηλαδή, τα κράτη-μέλη πρέπει να ξέρουν τι ακριβώ πρέπει να γίνει για να αλλάξουν οι πρακτικέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρια, Μάρια, συγγνώμη η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Όχι, δεν είναι η προηγούμενη εκπρόσωπος, αλλά ο κύριος Δεσιμονή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, όπως αναφέρει η αναφορά, το 2016 ήταν διάφοροι έλεγχοι, όχι προσωπικά δεν συμμετέσχουν, αλλά διάβασα τις ε, σχετικές εκθέσεις. Τα αποτελέσματα δείχνονται από ισορροπία, δεν υπάρχει συστηματικά καταστροφική κατάσταση και τώρα συντάσσουμε μια έκθεση, μια μελέτη όσον αφορά την κατάσταση και όταν ολοκληρωθεί η έκθεση θα την παρουσιάσουμε στα κρατημέλη τον Οκτώβριο και θα συζητούν τα κρατημέλη να πούν τι πιστεύουν, τι προοπτικές υπάρχουν και τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Κατά κάποιο τρόπο αυτό ακολούθησε αυτή την γενική άποψη, αυτή την προβληματική. Να δούμε πώς μπορούν να βελτιώσουν τα κανημερινή κατάσταση στο βαθμό που χρειάζεται. Θα πρέπει να δούμε προσοχή τα όσα εδώ αναφέρθηκαν γιατί είναι παλιά τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση. Τώρα, να προσθέσω αυτό που είπε προηγουμένως η Επιτροπή, ότι από τον Ιανουάριο έχουμε μια πλατφόρμα για την καλομεταχείριση των ζώων. Ξεκίνησε, θα ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου τις εργασίες της. Οπότε στην πλατφόρμα αυτή θα συναντώνται όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς να μπορούν να συζητήσουν και να δούμε πώς θα δοθεί κάποια συνέχεια στις καθημερινές αρχές που προβλέπονται για την μεταχείριση των ζώων σε κάθε τομέα. Σημαντικό είναι επίσης ότι έχουμε διαφορετικά αιτήματα. Δεν άρχισε βέβαια αυτή η Επιτροπή να εργάζεται, αλλά και εσείς, ίσως όχι εδώ, αλλά έχετε ψηφίσει για κουνέλια και για άλογα σχετικές εκθέσεις. Θα βάλουμε προτεραιότητες και η προσωπική μου γνώμη και εγώ της είναι ότι είναι πολύ καλός τομέας η γαλακτοφόρας γελάδες γιατί αφορά όλα τα κρατημένη. Πολλά αυτά τα ζώα. Έχουμε ένα σωρό επιστημονικά έργα σχετικά για τις σχετικές δραστηριότητες. Επομένως είναι σημαντικό να συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερομένους, να ενημερωθούμε στο πώς έχει η κατάσταση και να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα. Ο λόγος είναι για σας, κύριε Μάρια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κακομεταχείριση των ζώων και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Είδαμε από την αναφορά που την παρουσίασε ο αναφέρον την υπερεκμετάλλευση που γίνεται αυτή τη στιγμή στις γαλακτοφόρες αγελάδες, την κακομεταχείριση των ζώων αυτών, διότι ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή γάλακτος και έτσι να μεγιστοποιηθεί το κέρδος. Στις προηγούμενες όμως αναφορές είδαμε ότι οι τιμές του γάλακτος είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Είδαμε ότι η παραγωγή και ιδίως ε, όσοι έχουν, ε, εκτρέφουν αγελάδες ε, έχουν ένα χαμηλό εισόδημα. Ταυτόχρονα είδαμε να είναι ακριβές οι τιμές του γάλακτος σε σχέση με αυτά που πληρώνει ο καταναλωτής. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλη η κοινωνία έχει πει σε μια τεράστια αντίφαση. Κακομεταχείριση των ζώων, υπερεκμετάλλευση, αυξημένες τιμές για τους καταναλωτές, χαμηλό εισόδημα για τους παραγωγούς και προφανώς υπερκέρδη για τις επιχειρήσεις. Νομίζουμε λοιπόν ότι από την αναφορά αυτή είναι προφανές ότι η κοινωνία, η ευρωπαϊκή κοινωνία βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση και χρειάζεται, κυρία Πρόεδρος, άλλος δρόμος. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. And Peter now the floor is you. Äh, εγώ θα διατύπωνα την καταληκτική πρόταση με λίγο διαφορετικό τρόπο. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Το ζήτημα είναι αν είμαστε αρκετά γρήγοροι. Επειδή εγώ μεγάλωσα στο σοσιαλισμό. Εκεί είχαμε τη βιομηχανική γεωργία. Τότε, ως παράδειγμα το λέω, αν κοιτούσαμε στάβλους πριν από 40 χρόνια, τότε θα δείτε μόνο το 1 τέταρτο των ζώων πλέον βρίσκονται σε τέτοιε συνθήκε. Δηλαδή, όντω βελτιώσαμε πράγματα. Το ζήτημα είναι με ποια ταχύτητα. Εκεί έχει δίκιο ο κύριο Ματιά. Όλο αυτό πρέπει να γίνει στο κοινωνικό διάλογο. Τι είναι η ορθή μεταχείριση των ζώων, πώ την ορίζουμε, πώ την εφαρμόζουμε. Και πέρα από ένα πρακτικό οικονομικό ερώτημα, είναι οι όροι τους οποίους ε, θέλουμε να επιβάλλουμε σε όλη την Ευρώπη επειδή σε τελική ανάλυση είναι και όρια ανταγωνισμού. ανταγωνισμού. Γι' αυτό και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το ζήτημα αυτό και ο διάλογος πρέπει να λάβει χώρα. Επίσης όσον αφορά τους, τις συνθήκες και τους χρόνους μεταφοράς που, και άλλα ζητήματα που, που συζητούνται συχνά και στους τομείς αυτούς έχουμε, να κάνουμε, έχουμε έντονη αντίσταση από τα κράτη-μέλη, από κάποια κράτη-μέλη τουλάχιστον. Υπάρχουν διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, οπότε εγώ θα έλεγα το θέμα είναι σημαντικό. Η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή και πρέπει να αποσταλεί στις αρμόδιες επιτροπές ώστε να της δοθεί μια υποστηρικτική όθηση και οι επιτροπές να ασχοληθούν και πάλι με το ζήτημα. Επειδή εδώ παρουσιάζεται σαν να είναι οι οι κακοί που, που θέλουν να αποκτήσουν χρήματα από αλλά σε τελική ανάλυση είναι επιχειρηματίες επίσης. Πρέπει να επιβιώσουν οικονομικά και πρέπει να φροντίσουμε σε αυτό το πλαίσιο για καλές συνθήκες εκτροφής και ορθή μεταχείριση. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Μπορούμε να πούμε ότι αργούμε, αλλά δεν είναι ότι δεν γίνεται κάτι. Αν κοιτάξουμε τα πράγματα και συγκρίνουμε την κατάσταση με όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε κάτι για να δούμε πόσο αντιφατικά είναι τα συμφέροντα, πόσο αντικρουόμενα. Αφενός μαχηθήκαμε έντονα για την οδηγία για την οδηγία περί καθαρισμού με αποτέλε... θα... αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται τα βοηδή να εγκαταλείπουν τους στάβλους ποτέ και θα πρέπει να τους επιτρέπεται να εγκαταλείπουν τους στάβλους δηλαδή και να αφήνουν τα αέρια τους Οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε από τις αρμόδιες επιτροπές να ορίσουν κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή. Το, ζητού, το αντικείμενο δεν είναι μόνο οι αγελάδες, αλλά όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Αυτή είναι η υπεποίθησή μας. Πρέπει να σεβόμαστε τα πλάσματα στο πλανήτη μας, τα οποία ανήκουν και τα ζώα. Προτείνουμε δηλαδή να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή και να αποσταλεί στις αρμόδιες επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κανείς άλλο στον κατάλογο ομιλητών, οπότε ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Όχι, θα δώσουμε το λόγο στον αναφέροντα. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Κάτι να σχολιάσω. Στόσο είπε κάποια στιγμή για το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνα μας το 2012. Δεν νομίζω ότι και πολλά θα έχουν αλλάξει. Η δε έκθεση της DG Πολιτικές έγινε φέτος, στην αρχή του χρόνου. Αυτή η έκθεση έλεγε ότι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα μεταχείριση των ζώων, κακό μεταχείριση των ζώων είναι κακό μεταχείριση των γαλακτοφόρων αγελάδων. Και έχουμε αυτό το, την υπηρεσία Food and Veteran Office ε, με όλο το σεβασμό νομίζω ότι ε, παρά είναι ευγενική προς τον κλάδο για αυτά τα προβλήματα των γαλακτοφόρων αγελάδων. Πριν από δύο χρόνια απευθύναμε ένα ερωτηματολόγιο στα Υπουργεία Γεωργίας όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας πούν τι, τι, προβλήματα υπάρχουν, να μας πούν τι μπορεί να γίνει για την καλοδοχήση των αγελάδων. 12 ε, απήντησαν πάλι λέει αλλά περισσότερο περισσότερα κράτη-μέλη δεν είχαν ε, κάτσει να σκεφτούν τι θα πει το να κάνει κανείς να λάβει κανείς όλα τα λογικά μέτρα. Και είπαμε ότι θα βοηθούσε το να στείλει και ψενθεντήρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα πρόσφατα εξέδωσε τέτοιου είδους ε, καθοδίες, τέτοιες οδηγίες όσον αφορά την μεταφορά των ζών των ζώων. Και τα κρατη πρέπει να λάβουν τα σχετικά μέτρα και επίσης και οι αγρότες. Άρα χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιες κατευθυντήριες. Βοηθούν πολύ. Ε, ελπίζω η αναφορά μας να μείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα ε, λέγοντας ότι θα μείνει ανοιχτή η αναφορά και μετά τους, τους ελέγχους η Επιτροπή θα έχει πιο πλήρη εικόνα για το τι ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Οπότε μπορούν να ξανέλθουν εδώ και να μας τα εξηγήσουν. Άρα έχουμε αυτή την έκθεση των πέντε ελέγχων. Αυτά όλα θα πρέπει να ανελυθούν περισσότερο στην Επιτροπή μας. Και επίσης το τι θα γίνει με τη, στη συνάντηση του Οκτωβρίου στην Ιρλανδία. Θα πρέπει να ενημερωθούμε. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για την σημερινή κατάσταση στα κρατη και για το αν συμμορφώνονται με την οδηγία. Πολύ χρήσιμο. Άρα, περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο και να ξανέχουμε ανταλλαγή απόψεων για το ίδιο θέμα. Επίσης να στείλουμε επιστολή στην Επιτροπή Γεωργίας. Να τους ενημερώσουμε, να τους πούμε ότι ασχολούμεθα με το θέμα και ότι υπάρχει πρόοδος στη συνεργασία της Επιτροπής μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ναι, και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, λέει ο κύριος σωστά. Βλέπω γνέφη καταφατικά επιτροπή και αυτό με ικανοποιεί. Ωραία. Ελπίζω ότι σας ικανοποιεί η συζήτησή μας, λέω προς τον ε, αναφέροντα, μάλιστα μάλιστα. Οπότε ήμασταν χρήσιμοι για να πάρουν τα πράγματα τόσο στο δρόμο. Και ευχαριστούμε που κάνατε αυτό το ταξίδι για να έρθετε στις Βρυξέλλες. Α, σημερινή λιακάδα ελπίζω να σας δώσει ελπίδα που να τη φέρετε μαζί σα να την πάρετε μέσα στην πατρίδα σα. Και τώρα το τελευταίο μα θέμα για σήμερα είναι η Επιτροπή Εξεταστική Διευνητική στην Σουηδία που θα γίνει τον... που έγινε, που έγινε. Τον Φεβρουάριο, στην πατρίδα μου. Συνάδελφε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να σας πω σύντομα για την επίσκεψη του Φεβρουαρίου. Ήταν η επίσκεψη αυτή πολύ επιτυχής. Ποιο ήταν το θέμα. Οι Σουδικές αρχές για πάρα πολλές ταυτοποιήσεις που αφορούν αλλοδαπούς καθυστερούν καθυστερούν και έτσι καθυστερεί η συνολική διαδικασία που θα πρέπει να ισχύσει για αυτούς τους ε, αλλοδαπούς. Εμείς ήρθαμε σε συνεννόηση με τις Σουηδικές Αρχές. Συμφωνήσαμε για το πώς πρέπει να ενεργούν οι αρμόδιες αρχές. Που διατυπώσαμε κάποιες συστάσεις και από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία και από τις πολιτικές ομάδες, οπότε τον επόμενο μήνα θα ψηφίσουμε τη σχετική έκθεση. Το θέμα είναι βέβαια να ασχοληθεί κι άλλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Από ό,τι μαθαίνω, η σχετική αξιολόγηση δεν ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι οι Σουηδικές Αρχές στα λόγια. Ήταν πρόθυμες προς συνεργασία. Αλλά τα λόγια δεν τα ακολούθησαν έργα. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πιο αποφασιστικοί. Η προθεσμία για τις προπολογίες είναι 2 Μαΐου, στις 3 η ώρα. Thank you, Paul. Πάλι σε ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Λίγοι είχαν συμμετάσχει, αλλά τέλο πάντων ε, ας μα πούνε και οι άλλοι πώ τα είδαν τα πράγματα. Η κυρία Τζουφρίντα ευτυχώ είναι εδώ, αλλά και η κυρία Κούνεβα είναι εδώ. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Κυρία Τζουφρίντα πρώτη, ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, συμφωνώ. Ήταν χρήσιμη αυτή η αποστολή. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Αντιπρόεδρος ότι θα πρέπει αυτή η έκθεση να αποκτήσει περισσότερη πυγμή, να είναι πιο έντονη για να μπορέσουμε να πιέσουμε. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και ε, μέσα σε λίγο χρόνο πάρα πολύ ευχάριστο ήταν ότι κάναμε κάτι σαν επίδειξη δυνάμεων. Ε, μπορέσαμε επίσης να προσθέσουμε εμεί μέρα για να μπορέσουμε καλύτερα και εις βάθος να εξετάσουμε το πρόβλημα. Βέβαια συναντήσαμε ε, παντού ε, προθυμία από όλους τους ε, συνομιλητές μας για αυτό το θέμα που ξέρουμε ότι είναι τόσο σημαντικό και τελικά έγινε αντιληπτό ότι επήγε να βρεθεί μια λύση. Απόδειξη είναι ότι έχουμε όλες αυτές τις αναφορές. Έχουμε αναφορές που αφορούν διαφορετικές όψεις του προβλήματος και επίσης έχουμε λάβει τώρα κάποιες διαβεβαιώσεις μας ενημέρωσαν εξαντλητικά οι συνομιλητές μας και κάπου τα πήγαμε περισσότερο καλά από άλλα άλλα θέματα και θα πρέπει να δούμε για το ότι η σχέση των πολιτών με το Κοινοβούλιο με τέτοιες προσπάθειες συσφίγγεται. Άρα η Επιτροπή μας τελικά συμβάλλει στο να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε μια τέτοια περίοδο. Άρα και εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, θα πρέπει να προσέξουμε και να επιτευθεί ο στόχος αυτής της αποστολής, δηλαδή το να δούμε τι πάει στραβά με τις ειδικές αρχές. Να αποσπάσουμε δηλαδή κάποια από τα αποτελέσματα θετικά. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρχει τελικά ένας πάγιος διάλογος, να μην περιορίζεται μόνο στο χρονικό σημείο κατά το οποίο πάει μια κοινοβουλευτική ε, αποστολή στη χώρα που αφορούν τόσες και τόσες αναφορές οπότε τελικά δόθηκε άμεσα λύση ε, γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τι γίνεται και να προσέξουμε να ισχύουν στην πράξη τα δικαιώματα αυτών των ε, ανθρώπων, των νομίμως ε, κατοικούντων εκεί. Πολύ ενδιαφέρον επομένως να συμμετάσχουμε και βέβαια ευχαριστούμε την Πρόεδρο γιατί η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Ε, να ευχαριστήσουμε και τη γραμματεία μας και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν κάτι σαν κάτι ποστάλτο, πως, ε, πως εγώ από τον Νότο είδα την πόλη αυτή ντυμένη στα λευκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Κούνεβα, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο για τα επαναλαμβάνω όλες τις λεπτομέρειες. Θα πω κάποια πράγματα που με εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλά οργανωμένο το ταξίδι, ήταν πολύ καλή η ενημέρωση και από την κυβέρνηση και από τα υπουργεία, από τα γραφεία τα οποία ήδη είχαν ξεκινήσει και ασχολόταν με όλα τα θέματα που είχαμε θέσει από καιρό. Ε, έχουν πάρει πολύ σοβαρά τη ρύθμιση, η οποία βέβαια τα πάρει χρόνο. Α, το καλύτερο είναι ότι δεν έκαναν μόνο αυτά που χρειάζεται ε, από τους, ε, για τη ρύθμιση της νομοθεσίας επάνω στις αναφορές, αλλά είχαν ενταχθεί αλλαγή για να προσαρμόσουν έτσι τη νομοθεσία τους για να είναι ωφέλιμο και τους πρόσφυγες. Γιατί οι πρόσφυγες που πάνε από τα τελευταία χρόνια στη, Σουηδία έχουν τα ίδια ζητήματα. Έχουν ζητήματα με το προσωπικό αριθμό, έχουν ζητήματα με την πρόσβαση στις υπηρεσίες της χώρας. Και αυτό ήταν καλό. Από την άλλη πρέπει να συνεχίζουμε βέβαια για να παρακολουθούμε έως να ολοκληρώσει η διαδικασία, έως να εφαρμόσει όλες τις ρυθμίσεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την οργανωμένη επίσκεψη στη Σουηδία. Ήταν πολύ καλή. Well, I would simply like to, to highlight, I was there... Την πλευρά μου να πω ότι βεβαίω μια και είναι η χώρα από την οποία κατάγομαι ήμουν ε, παρούσα στην αποστολή εξοφίτσιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους που ήταν πολύ ουσιαστική στην, τη συνεισφορά τους στην επίλυση του προβλήματος. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την εξαιρετική οργάνωση της επίσκεψης. Νομίζω ότι απέδωσε ο καρπούς η επίσκεψή μας. Είμαι βέβαιη ότι οι αρχές του Σουηδία θα τα λάβουν τα θέματα αυτά σοβαρά. Δεν ε, συμβαίνει συχνά να λαμβάνουμε αναφορέ και να γίνονται και τέτοιου είδου επισκέψει στη Σουηδία. Επομένω, είναι σίγουρο ότι θα ληφθεί υπόψη σοβαρά. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Λου. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή και για την εξαιρετική έκθεση που ακολούθησε της επίσκεψης και η οποία περιγράφει το, το πρόβλημα με ακρίβεια. Όπως αναφέρεται, είμαστε ήδη σε επαφή με τις Σουηδικές Αρχές εδώ και καιρό και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε και διαδικασία pilot, πολιτική. Λάβαμε την απάντηση των Σουηδικών Αρχών το Φεβρουάριο, δηλαδή περίπου την ίδια περίοδο που εσείς οργανώσατε την Αποστολή σα ίσω αυτό να εξηγεί και την εξαιρετική προετοιμασία που είχαν να κάνει οι αρχέ τη Σουηδία, Η απάντηση που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ταιριάζει με τι πληροφορίε που έδωσαν οι Σουηδικέ αρχέ σε εσά. Αυτή τη στιγμή βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταλέξει στην τελική της θέση, περιμένουμε και τη μετάφραση ορισμένων αναγράφων, αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι ε, θεωρούμε την απάντηση αυτή ενδιαφέρουσα, αλλά παραμένουν ορισμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. Για παράδειγμα, οι λύσεις που προτείνουν οι Σουηδικές αρχές καλύπτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και το δεύτερο το οποίο σχετίζεται και με αυτό που ανέφεραν οι βουλευτές, θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι σουηδικές αρχές ότι υφίσταται η πολιτική βούληση για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και η πολιτική βούληση για να υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υποσχέσεις. Αλλά δεν αρκεί. Ε, σίγουρα δεν θα αρκούσε αυτό για να κλείσουμε την πιλωτική υπόθεση που ανοίξαμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία μας με τις Σουηδικές Αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ζητεί κάποιος άλλο συνάδελφος τον λόγο για να προσθέσει κάτι. Ίσως ο υπεύθυνο της επικεφαλής της αποστολής. Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Θα συνεχιστεί η παρακολούθηση της υπόθεσης από την Επιτροπή. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα μας ενημερώσετε θα ενημερώνεται το κοινοβούλιο δηλαδή. Πάντω, σίγουρα μπορώ να σα πω ω Σουηδέζα, ότι ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν ιερό για εμά. Είναι, μια ε, νοτροπία που υπάρχει, αλλά πρέπει να, πρέπει να αλλάξει, γιατί δημιουργεί στην ουσία διακρίσεις και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Προθεσμία τροπολογιών 2 Μαΐου, 3 μετά μεσημβρίαν, ε, οι τροπολογίε μπορούν να αφορούν μόνο στις συστάσεις. Η ψηφοφορία θα γίνει 30 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε αύριο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.